διάσκεψη. Κλείνει λοιπόν η συζήτηση, λίγη η συζήτηση. Επαναλαμβάνω ότι έλαβα έξι προτάσεις ψηφίσματος. Η συζήτηση έχει λήξει και περνάμε στην ψηφοφορία. Αρχίζουμε με το ΣΥΝΑ, με την παράνομη διακίνηση ανθρώπων στο ΣΥΝΑ. Παράγραφος 4, τροπολογία 3, ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στο αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ε, αποχές με συγχωρείτε δεν το είπα, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές ε, επαλήθευση δεν είμαστε σίγουροι. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά υπέρ. Α, με συγχωρείτε, αρχίζει η ψηφοφορία, λέει πρόεδρος, πέρας. Απορρίπτεται. Πέντε υπέρ. Ένα, Με συγχωρείτε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην Παλαιστίνη, στις επιδρομές των Ισραηλινών δυνάμεων σε Παλαιστινιακούς σταθμούς. Σύνολο λοιπόν της πρότασης υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στο τρίτο κείμενο στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δύο. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρία. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το αρχικό κείμενο. 10, εδάφιο 10 του αρχικού κειμένου. Όχι, με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος, υπάρχει μία προφορική του Τάνοκ, του κυρίου Τάνοκ. Ποιος είναι υπέρ του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί. Ο κύριος Τάνοκ δεν είναι παρόν. Θα ήθελε κάποιος να αιτιολογήσει. Εντάξει, περνάμε στο 1 κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία και αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Έτσι λήγουν οι σημερινές μας εργασίες. Ε, μία πληροφόρηση και μόνο από το ΕΛΚ ζητήθηκε στην, στον έλεγχο προϋπολεσμού η κυρία Πέτρη Σαρβάμα, το ίδιο στην Επιτροπή Μεταφορών και στη συνεργασία Μικτή Επιτροπή